συνάδελφοι και συναδέλφισες επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση τα πρακτικά της χθεσινής ε, συνεδρίασης ε, είναι στην διάθεσή σας υπάρχουν αντιρρήσεις αντίρρηση ή θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο μάλιστα πείτε μας ωραία λοιπόν αντιρρήσεις δεν υπάρχουν ε? ή όχι είναι αντιρρήσεις τελικά Α, να του δώσω το λόγο. Εκεί στο 839. Α, και έτσι διάει. Α, δεν έχετε αντιρρήσει για τα πρακτικά. Εγκρίνονται λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, δήλωση της Κομισιόν για τις συστάσεις ε, για το άνοιγμα διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ και χαίρομαι που καλωσορίζω την Επίτροπο, την κυρία Μάλμστρομ. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, η κοινή συμφωνία μεταξύ των Πρόεδρων Γιούνκερ και Τραμπ του περασμένου Ιουλίου παρουσίασε μια θετική εμπορική ατζέντα με τι ΗΠΑ το πιο σημαντικό μα εμπορικό εταίρο και βοήθησε στο να αποκλιμακωθούν οι εντάσει ε, με αυτή την πολύ κρίσιμη σχέση. Από τον περασμένο Ιούλιο συνάντησα ε, πέντε φορές ε, τον ομόλογό μου για να αναθεωρήσουμε την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας ε, και να εντοπίσουμε την κοινή δήλωση. Την περασμένη εβδομάδα στη συνάντησή μας αξιολογήσαμε την πρόοδο στα διάφορες εργασίες και τον ενημέρωσα για την διαδικασία υιοθέτηση των εγκρίσεων διαπραγματεύσεις. Του είπα ότι στο Συμβούλιο θα ολοκληρώσουμε τις συζητήσει ε, για τις εγκρίσεις ε, και για την εξάλληψη των δασμών για τα ε, βιομηχανή προϊόντα και το άλλο για την αξιολόγηση συμμορφωσης και περιμένω να γίνει σεβαστή εφαρμογή της κοινή δήλωση όσο έχει και ότι οι μελλοντικέ διαπραγματεύσεις δεν θα θίξουν την αργία. Είμαι σίγουρη ότι ο οίκος σας γνωρίζει πόσο σημαντικές είναι οι αδιαδηλαντικέ εμπορικές σχέσεις που ήταν και θα μείνουν κεντρική αρτηρία τη παγκόσμια οικονομίας ε, μια ε, ατζέντα που θα έχει σχεδιαστεί σωστά μπορεί να μας ωφελήσει όλους. Δεδομένου του μέγεθος των εμπορικών σχέσεων, η εξάλληψη των δασμών, ακόμη και αν σήμερα είναι σχετικά χαμηλή, οδηγεί σε σημαντική μείωση του κόστους ε, για τους παγκόσμιους οικονομικούς φορείς. Πολλοί βιομηχανικοί τομείς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ε, λειτουργούν ε, με μικρά περιθώρια κέρδους λόγω της αποτελεσματικότητας των αγορών μας. Μία περιορισμένη συμφωνία για τα βιομηχά αγαθά και τους δεσμούς θα έδινε στις διατλαντικές εταιρείες όλων των μεγεθών συγκριτικό πλεονέκτημα και θα υποστηρίζει την παγκόσμια ικανότητά του να ανταγωνιστούν. Εμεί εκτιμούμε ότι θα υπάρχει ε, αυξημένη ε, ε, περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση κατά 8% στις εμπορικές συναλλαγές και εργάζομαι και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης θα μπορούσαμε να έχουμε οικονομικά ωφέλη για μια συμφωνία ελευθεροπορία για τα βιομηχανικά προϊόντα. Ξεκινήσαμε τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφέρομενα μέρη την περασμένη εβδομάδα και τους καλέσαμε να εξετάσουν τις προτάσεις μας και περιμένουμε να λάβουμε την υποστήριξή τους για τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ στον τομέα αυτό. Γνωρίζω ότι κάποιοι εξημών φοβούνται ότι θα διαπραγματευτούμε υπό απειλή και θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω ότι έχω στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους εταίρους μας την ε, περασμένη εβδομάδα αλλά και πιο πριν ότι οι μονομερεί εμπορικέ δράσει από τι Ηνωμένες για τι εισαγωγέ ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν ε, να προκαλέσουν ζημία στι σχέσει μα σε κρίσιμη στιγμή. Επίση, ε, του είπα ότι δεν θα το επιλέξουμε αν λάβει μονομερή μέτρα η Αμερική. εμεί θα απαντήσουμε αμέσω, θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσει αμέσω και αυτό προβλέπεται ξεκάθαρα στο σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών και επίση θα υιοθετήσουμε μέτρα εξισορρόπηση. Βέβαια ελπίζουμε ότι η λογική θα υπερισχύσει και δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την οικοδόμηση τη σχέση αυτή με ε, επωφελή αποτελέσματα και για του δύο. Η έγκαιρη υιοθέτηση αυτών των εντολών θα είναι σημαντικό μήνυμα της καλής πίστης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, να τιμήσει τι δηλώσει του περασμένου Ιουλίου. Η καθυστέρηση ε, στην ε, υιοθέτηση ε, έχει οδηγήσει σε λαθασμένου ισχυρισμού για τη δέσμευση των ΗΠΑ. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υποστηρίξετε τι διαπραγματεύσει μα με τι ΗΠΑ. Η σημασία τη δική σα υποστήριξη είναι πολύ μεγάλη. Θα δείξει ενότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ενότητα είναι η δύναμή μα. Σε αντίθεση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια ψηφοφορία από το Κοινοβούλιο κατά αυτών των ε, περιορισμένων διαπραγματεύσεων θα ήταν μια ψήφο κατά μια καλά ισορροπημένη και αναλογική προσέγγιση τη δήλωση του Ιουλίου που αναπτύξαμε για να μειώσουμε τι εμπορικέ εντάσει. Επομένω, ε, θα υπερψηφίσετε για να διατηρήσετε τι σημερινέ εντάσει με τι Ηνωμένε ενώ Έχουμε ιδέε για να μειώσουμε τι εντάσει αυτέ αυτή τη στιγμή επιτάπητο. Και σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, καθώ τα έχουμε συμπεριλάβει στην πρότασή μα, είναι πολύ καλύτερο για την ε, διατλαντική σχέση να μειωθούν οι δασμοί στα αυτοκίνητα στο 0%. Είναι καλύτερο για τους παραγωγούς, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές. Πολύ καλύτερο από το να έχουμε περαιτέρω δασμού στα αυτοκίνητα και στα εξαρτήματα. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τις ε, δικές σας σκέψεις ε, και τις συστάσεις σας και να επαναλάβω ότι μόλις θα έχουμε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις θα ενημερώνουμε αυτό τον οίκο για όλε τι στοιχείες των συζητήσεων, όπως κάνουμε πάντα για τα εμπορικά ζητήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Äh, Σα ευχαριστώ. Τώρα ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματο των εισηγητών. Για το ΕΛΚ, η κυρία Κβίστχαουτ Ρόβολ. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω τον σεβασμό μου στις προσπάθειές σας να ομαλοποιήσετε ξανά την διατλαντική σχέση. Και μόνο μέσω επικοδομητικών συνομιλιών θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό ελπίζω να σας ενθαρρύνει αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας δώσει μια τέτοια εντολή. Είναι προς το συμφέρον όλων μας να εξερευνήσουμε πιθανά κοινά σημεία με τις είπα για να πέσει η ένταση στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως, ε, αυτοί οι οποίοι λένε πως μόνο σκληρή γρόσα καταλαβαίνει ο Τραμπ, ε, ίσως δεν είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν την καθημερινή και φέρνουν την καθημερινή ζημιά είτε στον τομέα των αυτοκινήτων είτε σε άλλους κλάδους. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουν ΙΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν έχουμε και να χάσουμε τίποτα. Εάν δεν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον θα έχουμε κάνει μία προσπάθεια. Αν έχουν αποτέλεσμα, δεν θα έχουμε απλώς παραμερίσει την εμπορική διαφορά, αλλά και τους δασμούς και τα εμπόδια στο εμπόριο. Και τέλος, να πω μία λέξη ακόμα. Ο κόσμος κινείται, προχωράει. Μα εμείς διαπραγματευτούμε Τι διαπραγματευτούμε, αυτά συμβαίνουν. Και πρέπει οι μεγάλες δημοκρατίες να συνεργαστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κύριε Λάγκε, έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Δεν θα διαπραγματευτούμε με το όπλο στον κροταφό. Αυτό το ακούσαμε σε πολλές δηλώσεις τις τελευταίες μέρες. Ότι δεν θα διαπραγματευτούμε εκβιαζόμενοι. Και τώρα αναρωτιέμαι τι άλλαξε. Οι δασμοί των ΙΠΑ σε χάλιβα και αλουμίνιο εξακολουθούν να ισχύουν. Υπάρχουν και άλλοι δασμοί στο, ε, στις ισπανικές Έχουμε την απειλή του Τραμπ για επιπρόσθετους συντασμούς στα αυτοκίνητα και στα ανταλλακτικά. Δεδομένης της, είπας, ε, της, ε, της πίεσης των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τι συνέβη λοιπόν. Έχουμε κάνει εμείς υποχωρήσεις. 180% αύξηση των ε, εισαγωγών ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης ανάλογη αύξηση ε, σόγιας, των εισαγωγών σόγιας από τις ΗΠΑ τα οποία μετά αναμειγνύονται στο βιοδίζελ. Κι άλλη δηλαδή αύξηση των εισαγωγών αυτών. Λοιπόν, έχουμε κάνει και παραχωρήσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι οι παραχωρήσεις των ΗΠΑ έχει πέσει καθόλου η πίεση των είπα, Εγώ δεν βλέπω τίποτα τέτοιο. Και όσο ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να διατυπώσουμε την θέση μας με αυτοποίηση. Δεύτερον, τον Ιούλιο πέρσι, αγαπητοί συνάδελφοι, αποφασίσαμε να μην κλείσουμε συμφωνία χωρίς αναφορά στην Συμφωνία των Παρισίων. Σήμερα, λίγες ώρες πριν από αυτήν την συζήτηση, συζητούσαμε για την προστασία του κλίματος. Όλα αυτά δεν υπάρχουν στην διαπραγματευτική εντολή. Τίποτα. Ούτε μία αξιολόγηση αντικτύπου. Όχι. Πρέπει να διατυπώσουμε τις απαιτήσει μας. Πρέπει να απορρίψουμε το δίκαιο του ισχυρού και να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τους κανόνες. Σας ευχαριστώ για το ECR. Έχει τον λόγο ο κύριος Ζάχραντιλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, η διατραντική εταιρική σχέση είναι ο λίθος του του συστήματός μα και στηρίζουμε αυτή την πρόταση για τους δασμούς για τα ε, βιομηχανικά αγαθά και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Αυτό θα φέρει σημαντικά ωφέλη στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, ε, η κατάργηση των υψηλών δασμών στα μεταποιημένα προϊόντα όπως είναι τα ε, διένδυση και υπόδηση θα ανοίξει ευκαιρίες για εξαγωγής ε, και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας. Επιπρόσθετα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποφεληθούν από την επικάλυψη ε, των δοκιμών και των πιστοποιήσεων σύμφωνα με την αξιολογική της Θα ήθελα να προσθέσω έναν όρο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ότι δεν μπορούν να ε, κλείσουν επιτυχώς χωρίς ε, την άρση των δασμών στον χάλιβα και το αλουμίνιο. Χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια για τον, τη συμπερίληψη του τομέα του αυτοκινήτου ε, έτσι ώστε να υπάρχει ε, συμμόρφωση με τους κανόνες ε, του ΠΟΕ και πιστεύω ότι είπα και οι ΕΕ θα πρέπει να μάθουν μετά από τις διαπραγματεύσεις της TTIP ιδιαίτερα για θέματα δασμών, διευκολύνσεων τελωνιακών και η ομάδα μας ελπίζει ότι αυτό θα αποτελέσει τη βάση για περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο τη άλλη, κυρία Σχάκη, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Το εμπόριο με βάση τους κανόνες είναι σημαντικό για τις οικονομίες μας, ειδικά καθώς η ανάπτυξη της επόμενης δεκαετίας θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτώντας την Κίνα βλέπουμε μια χώρα η οποία δεν σέβεται του εμπορικού κανόνε και δυστυχώ και στις ΗΠΑ βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει θεωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απειλή για την εθνική ασφάλεια για να δικαιολογήσει τους δασμούς της και εντωμεταξύ βεβαίως μας υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις μας στο ΝΑΤΟ. Ε, δεν στέκουν αυτά και η κλιμάκωση των ε, σχέσεών μας θα έχει σοβαρές συνέπειες. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να συνομιλούμε και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Κάποιος πρέπει να είναι ο ενήλικος στην αίθουσα. Οπότε, για αυτούς που δεν θέλουν να στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζω να αντιλαμβάνεστε, θα σας τα εξηγήσει και ο πρέσβης, ο κ. Σάντερλαντ και οι υπόλοιποι, ότι αυτά θα θεωρηθούν απόδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι ανίκανη να λαμβάνει αποφάσεις. Λοιπόν, δεν πρέπει να εμποδίσουμε την ε, έναρξη διαπραγματεύσεων με περιορισμένη ε, βάση. Δεν μιλάμε για ξεπάγωμα τη TTIP με το να υποστηρίξουμε το άνοιγμα αυτών των διαπραγματεύσεων αλλά υπό πολύ συγκεκριμένου όρου πριν ολοκληρωθούν αυτέ έχουμε κάποιε διαπραγματεύσει που έχουν νόημα. Θα ήθελα επίση να πω σε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι συμφωνίε με τρίτε χώρε ω ένα εργαλείο για να πλήξουν αυτέ τι χώρε ενώ δεν έχουμε τα θεμέλια διμερών συμφωνιών ε, με τις χώρες με τις οποίες κάνουμε εμπόριο, όπως η Κίνα. Οπότε σκεφτούμε τι έχουμε να κερδίσουμε, αλλά και το τι έχουμε να χάσουμε εδώ πέρα. Οπότε η ομάδα μου στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ισχυροί και ενωμένοι ως Ευρώπη. Ειδικά όταν ε, αντιμετωπίζουμε την κυβέρνηση Τραμπ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για τους ε, πράσινους, ο κύριος Ζαντό για δύο λεπτά. Κυρία Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Ντόναλτ Τραμπ είναι αυτός που πριν από κάποια χρόνια έλεγε ότι η κλιματική αλλαγή είναι μεγάλη απάτη. Είναι μια έννοια που έχει εφευρεθεί από και για τους Κινέζους προκειμένου να κάνουν μια ανταγωνιστική την μεταπητική βιομηχανία. Και όταν το Κογκρέσο έκανε μια έκθεση 300 επιστήμονες έλεγαν ότι η κλιματική αλλαγή είναι δραματική και για τις ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ έλεγε δεν το πιστεύω. Αυτός ο ίδιος, ο πρόεδρος Τραμπ, τους τελευταίους μήνες δεν έχει σταματήσει ε, να υποδαβλίζει το Brexit, υποστηρίζει το πιο σκληρό Brexit και μάλιστα και κριτική και στην Τερέζα Μέη για τη βούλησή της να βρει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με τον πρόεδρο αυτό είναι που θέλετε σήμερα να διαπραγματευτείτε είναι με τον πρόεδρο αυτό, στον πρόεδρο αυτό που δίνεται ένα μέρος της ε, κυριαρχίας μας και των αξιών μας. Έχει υποθεί αυτό, το είπαν ε, και οι σοσιαλδημοκράτες ε, φίλοι μας έχουν βρει μάλιστα τη λογική σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Δεν διαπραγματευόμαστε με ένα πρόεδρο που μας θέτει το πιστόλι στον κρόταφο. Δεν διαπραγματευόμαστε με έναν πρόεδρο που ε, μας ε, απειλεί για τα αυτοκίνητα, ε, για την συντηρουργία και μας θέτει και φόρους. Είναι μια πολιτική και οικονομική δύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλετε να το δείξετε αυτό, και αν θέλετε να δείξουμε ότι περασπίζουμε τις αξίες μας για το κλίμα και για τα κοινωνικά και και περιβαλλοντικά ζητήματα, τότε δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, γιατί είναι γελίο να θεωρούμε ότι θα ξεκινήσουμε και κατόπιν θα δούμε στην πορεία. Όχι, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε σήμερα με τις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί ο πρόεδρος αυτός δεν εκπροσωπεί τις αξίες μας, ούτε τις ενσαρκώνει, αποτελεί κίνδυνο για την οικονομική μας κυριαρχία και τη δημοκρατική μας κυριαρχία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς, εξ ονόματος της Γκουέ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, κυρία Μάλμστρομ. Ο Πρόεδρος Τραμπ μας απειλεί και λέει θα σας ταράξω στους δασμούς. Τι να σου πω, δηλαδή αυτά ακούγονται σαν western. Εσείς είπατε πριν από ένα χρόνο ότι θα διαπραγματευτούμε μόνο όταν βγάλει τον πιστόλι από το τραπέζι ο Τραμπ. Και τώρα παραδίνεστε. Παρά την αυξημένη πίεση με τιμωρητικού δασμούς. Και μάλιστα παραβιάζεται και τις ίδιε σας τις αρχές, παρά το ότι η ουσιαστική συμφωνία αφορά πάνω από 90% των αγαθών τα οποία εμπορευόμαστε με τις ΗΠΑ, αρνείστε να γίνει μια ε, αξιολόγηση αντικτύπου οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει καμία διαβούλευση. Επιπλέον, έχετε κλείσει τα αυτιά και κάνετε ότι δεν ακούτε ότι ο Τραμπ είπε ότι θα εγκαταλείψει την συμφωνία των ε, Παρισίων. Εμείς θεωρούμε ότι έχει αποκλείσει εαυτόν η κυβέρνηση Τραμπ ως ε, διαπραγματευτικός εταίρος. Βεβαίως, το να υποκύψουμε εδώ πέρα θα σήμαινε το τέλος ε, και για χιλιάδες αγρότες μας. Ε, έχετε ξεχάσει την αντίδραση χιλιάδων εκατομμυρίων Ευρωπαίων στην ε, TTIP. Κυρία Επίτροπε, εγώ θα ζητήσω με τις τροπολογίες μας αύριο να μην σας δοθεί διαπραγματευτική εντολή από το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ για το EFTT η κυρία Μπεγιάν. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η θέση μα για αυτή τη δεύτερη εκδοχή τη TTIP δεν έχει αλλάξει, αλλά αυτή τη Επιτροπή, από ό,τι φαίνεται, ναι. Δεδομένου ότι από αμερικανικέ πηγέ η Γεωργία θα συμπεριληφθεί στη συμφωνία. Είναι βέβαιο, το ξέρουμε, γιατί ανοίγει την όρεξη στου Αμερικανού. Όμω, ε, ε, δεν είμαστε εμεί αυτοί που πρέπει να τηρούμε τη χείρα στι ΗΠΑ. Εμεί κάναμε ήδη αυτό που μα αναλογούσε, εισαγώντα το 75% τη δική του όγια και το 181% του φυσικού του αερίου. Τώρα είναι η στιγμή που αυτοί πρέπει να έρθουν να μας συναντήσουν. Πριν να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, θα θέλαμε η κυβέρνηση τον είπα να διακόψει τους δασμούς ε, για το αλουμίνιο και το χάλιβα και να διακόψει κάθε εχθρική πράξη κατά των αυτοκινήτων μας. Θέλουμε μια νέα συμφωνία, πολύ ωραία, αλλά ας ακυρώσουμε τη διαπραγματευτική εντολή της παλιάς συμφωνίας, ας ξεκινήσουμε το μηδέν και ας ακυρώσουμε για πάντα την που, που τρομοκράτησε για χρόνια τους Ευρωπαίους πολίτες. Και σας παρακαλώ να μην ξεπουλήσουμε τη γεωργία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι. Αυτό το ψήφισμα είναι περίεργο. Το πνεύμα του κειμένου έχει αλλάξει ε, και αποτελείται από ε, κείμενα του, της Άλτε, των ΕΛΚ, γιατί κάποιοι συνάδελφοι έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ε, ορισμένες αξίες. Ε, θα πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις εγγυήσει απέναντι στις είπε πριν αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Τώρα θέλουμε να διαπραγματευτούμε πριν να έχουμε τις βάσιμες και γερές εγγυήσει για τον τομέα του αυτοκινήτου, για την κλεισμό της γεωργίας πριν από τις διαπραγματεύσεις και σε ένα σύμφωνο που αφορά τον τομέα της αλίας. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι μια τέτοια συμφωνία ε, δεν θα υπογραφεί εάν οι συνθήκε δεν πληρούνται στο τέλο των διαπραγματεύσεων. Κανεί θα πρέπει απαραίτητα να θέσουμε του όρους μα στις ΗΠΑ πριν καθίσουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και σίγουρα όχι το αντίθετο. Σα ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στους συναδέλφου. Ε, που μιλούν ε, εξ ονόματο του κ. Η Επιτροπή Juncker έπρεπε να διορθώσει την ε, εμπορική πολιτική μετά από την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσυρθούν από την TTIP. Η αλήθεια είναι ότι οι κυρώσει για το αλουμίνιο και το χάλιβα θα πρέπει να εξελιχθούν όπω και για τι ισπανικέ ελιέ και δεν είναι η καλύτερη αρχή. Η δήλωση του περασμένου Ιουλίου και αυτέ οι διαπραγματευτικέ οδηγίε για την ε, μείωση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα και για του δασμολογικού φραγμού είναι κατά ενδιαφέρον όμως, Επίτροπε, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τις αρχές. Ε, βέβαια, πολλοί αναφέρονται στις αρχές της εμπορική μας πολιτική, όταν δεν πιστεύουν ούτε πίστεψαν και το χρησιμοποιούν ω πρόφαση για να απορριφθούν συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών. Είναι σημαντικό να αγωνιστούμε για ένα εμπόριο που θα βασίζεται σε κανόνε για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, να διατηρήσουμε τι αρχέ του Παρισιού και κυρίω να μην αγκαταλείψουμε τι ε, συμφωνίε που έχουμε με τη Μερκοσούρ, ε, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Μποστινάρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, όλοι συμφωνούμε εδώ ότι οι διατλαντικές σχέσεις ε, αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις ε, και αναταραχές ε, σε μικρό χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά είμαι πεπισμένος ότι ε, παραμένουν ε, ε, μακροπρόθεσμα θεμελιώδεις αξίες. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέτρα για να προστατεύσει την εσωτερική αγορά, τις βιομηχανίες και τους εργαζόμενους μας. Δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ γρήγορα οποιασδήποτε νέους δεσμούς και μέτρα λάβει η Αμερικανική κυβέρνηση. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να μειώσουμε τις εντάσεις και να αποφύγουμε την κλιμάκωση ενός εμπορικού πολέμου γιατί θα είναι οι συνέπειες μεγάλες και για τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε νέους δεσμούς παρά ο διάλογος και διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό εμπιστεύομαι η Κομισιόν θα κάνει το σωστό και καλωσορίζω τις προσπάθειες του Πρόεδρου Γιούνκερ και της Επιτρόπου Μάλστρομ και υποστηρίζω να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες για περιορισμένες τομέκες διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Και θα κλείσω με μια ερώτηση, κύριε Επίτροπε. Αν πούμε όχι στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ποιον λέμε ναι στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Χαρανσόβα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, η ΕΠΑ ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα φυσική εταίροι Έχουμε κοινέ αξίες και αντιμετωπίζουμε κοινέ απειλέ. Σε οποιαδήποτε σχέση βεβαίω υπάρχουν και τα δύσκολα. Παρά τα εμπόδια, τα θεμελιώδη κοινά συμφέροντα της ε, σχέσης μας είναι ισχυρά. Πέρσι είχαμε σαφώς ένα ιστορικό χαμηλό Αντιδρώντας ε, στους δασμούς για χάλιβα και αλουμίνιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ταυτόχρονα ότι είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί και το μήνυμα ήταν σαφές. Πρέπει να συνεργαστούμε. Το χρειαζόμαστε αυτό για τις επιχειρήσεις μας, ε, για τις δουλειές που δημιουργούν στην Ευρώπη. Οι αγορές μας, οι πόροι, η ασφάλεια και οι πολίτες μας ε, είναι αλληλοεξαρτώμενα και θα συνεχίσει αυτό να είναι έτσι στο μέλλον. Οπότε ελπίζω το κοινοβούλιο αυτό θα στηρίξει πλήρως την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Πάντα κερδίζουμε και μπορούμε να κερδίσουμε από τις διαπραγματεύσεις, αλλά αν κλείσουμε την πόρτα είπα, μόνο θα χάσουμε. Σας ευχαριστώ. Beauty Coffer για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, αγαπητοί συναδελφοί, η επίσκεψη του Πρόεδρου Γιούνκερ τον Ιούλιο ήταν μεγαλοφύης. Εάν η Κομισιόν είχε υποβάλει γρήγορα τότε ένα σχέδιο εντολής θα τα είχαμε ήδη καταφέρει. Αλλά δυστυχώς ξόδεψε χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο και οδηγηθήκαμε έτσι σε μια δημόσια συζήτηση και σε μια υποτίμηση της επιμονής της Αμερικανικής κυβέρνησης. Είπατε η ίδια ότι μονομερείς δράσεις θα βλάψουν τις διατλαντικές σχέσεις μας. Ναι, έτσι μιλάνε όσοι φοβούνται. Ο κύριος Λάιτάιζερ μας διατάζει από την άλλη. Και είναι πάρα πολύ απλά. Αν συμπεριφέρεται κανείς με την ουρά στα σκέλια, θα συνεχίσει να τρώει φάπες. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να απορρίψουμε αυτή την εντολή, να επανέλθετε και να μας υποβάλλετε μια καλύτερη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σάντσες Καλδεντά, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε για την κλιματική αλλαγή και η δεξιά γεμίσε το στόμα τη ε, με κενά λόγια μέχρι και ο Επίτροπο Κανιέται ήταν ανήσυχο για το μέλλον του πλανήτη. Λέω ότι δεν θα είναι τόσο εσεί ε, όταν ε, την Γκρέτα Τούμπερκ την απαγορεύσατε στα 10 και ήταν μόνο 16 ετών. Φοβάστε να ακούσετε την αλήθεια η πλευσία των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, ε, προωθούν τη δυναμική επιτάχυνση ε, τη κλιματική αλλαγή. Και εδώ έχουμε το παράδειγμα ότι αναβιώνουμε την TTIP, τη ανάτζεται όνομα και πιστεύω ότι θα περάσει αυτό χωρί να το καταλάβει κανεί. Κυρία Μάστροπ, δεσμευτήκατε ότι θα ήταν απαραίτητη η προπόθεση η εφαρμογή τη Συμφωνία των Περισσίων για την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών. Όλοι ξέρουμε τι σκέφτεται ο Τραμπ για την κλιματική αλλαγή και ότι αρνείται τη συμφωνία. Όμω οι επιχειρήσει είναι επιχειρήσει και αυτό έχει μεγαλύτερο βάρο από το μέλλον του πλανήτη. Ε, καθώ έχουμε νικήσει μια φορά την TTIP, ξέρουμε πω να το κάνουμε με ενημέρωση και κινητοποιήσουμε σήμερα. Υπάρχει και μια νεολαία που έχει ξεσηκωθεί και με ένα φεμινιστικό κίνημα δεν θα επιτρέψουν να προχωρήσουν πολιτικέ που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον μα Χρειαζόμαστε άλλο εμπορικό μοντέλο και θα το κάνουμε ενώ προλαβαίνουμε. Ευχαριστώ κύριε Ντάτμουθ, ένα μισή λεπτό. Uh, ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες ε, εξάγουν, εξήγαγαν αυτοκίνητα στη τιμή των 20 δισεκατομμυρίων το 2017. Και αυτό παρά το γεγονό ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίε είχαν ε, λίγη ε, εμπλοκή στην, στην στο να κανονίσουν τους Τώρα, οι δασμοί στα εισαγόμενα αυτοκίνητα ε, μέχρι 1,5%. Οι ευρωπαϊκή δασμοί σε αυτοκίνητα που εξάγονται από τις ΗΠΑ είναι 10%. Είναι ασύμετρο αυτό. Η Αμερικανική ε, διοίκηση έχει ε, κάτι να πει. Ό,τι και να λένε οι συνάδελφοι. Και ω αποτέλεσμα, οι εξαγωγέ αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μικρό κλάσμα. Μόνο 48 εκατομμύρια δολάρια έναντι 20 ε, δι. Τώρα, το ψήφισμα. Το ψήφισμα επικρίνει τη ΕΠΑ και την αποχώρηση από την Συμφωνία των Παρισιών. Αλλά κύριε Ζαντό, δεν μπορείτε να έχετε την κυβέρνηση που έχετε στην χώρα κάποιανού άλλου. Δεν μπορείτε να έχετε την κυβέρνηση που έχετε ούτε και στη δικιά σας χώρα. Το ξέρω εγώ αυτό πολύ καλά και το ξέρω και χρόνια. Τώρα, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ναι, είναι η πολιτικοποίηση του εμπορίου. Η πολιτικοποίηση ε, όλη αυτή στο ψήφισμα δείχνει πόσο δύσκολο είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση να οριστικοποιήσει αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Και αυτό, αυτές είναι οι κυρώσεις που πρέπει να πληρώσουν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτικοποίηση του ε, εμπορίου που υποβοηθείται από τόσους ε, πολλούς από εμά συναδέλφους. Σας παρακαλώ. Ναι. Ε, έχετε μια μπλε κάρτα. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Συνάδελφε, δεν κατάλαβα ακριβώ αν είστε πεπισμένο για την απορρίθμιση του κλίματο ή αν δεν είστε πεπισμένο για την απορρίθμιση του κλίματο. Δεν το κατάλαβα. Εάν η ε, Μεγάλη Βρετανία, που είναι μια μεγάλη χώρα στην ε, διεθνή κοινότητα, πίστευε πάντα στι ε, ανθρώπινε αξίε αυτή τη διεθνού κοινότητα. Και δεν κατάλαβα επίση εάν η κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα, αυτή τη στιγμή τη ψηφοφορία, είναι η δική σα κυβέρνηση. Δύο είναι αυτέ οι ερωτήσει. Θα απαντήσω τη μία, εάν δεν σας πειράζει. Στην συζήτηση αυτή συζητάμε το εμπόριο, όχι την κλιματική αλλαγή. Και είναι σοβαρό αυτό το οποίο λέω. Ότι πολύ απλά δεν πρέπει να κολλάμε άσχετα πράγματα περί κλιματικής αλλαγής και άλλα άσχετα. Ότι την πολιτική σας πείρα, τα ξέρετε αυτά, σε πολύ απλές εμπορικές συμφωνίες. Αν το κάνετε αυτό θα κοστίσει στους ανθρώπους της Ευρώπης, στους οποίους λέτε ότι εκπροσωπείτε. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Χάνσεν. Ευχαριστώ. Οι εμπορικέ συγκρούσει ξεκινούν όταν μια χώρα αποφασίζει να παραβιάσει του διεθνεί παραβιά κανόνε ε, για να ζημιώσει τι βιομηχανίε άλλων χωρών. Ακριβώ έτσι έχουν οι σχέσει μα με τι ΗΠΑ. Ο στόχο μα θα πρέπει να είναι να είμαστε ισχυροί για να προωθήσουμε τι εξαγωγέ μα. Όσοι προσπαθούν να δορπολίσουν στι διαπραγματεύσει με τι ε, ΗΠΑ τελικά διακινδυνεύουν τι θέσει εργασία ε, του λαού. Το 88% των ευρωπαϊκών εταιριών που εξέγουν στι ΗΠΑ είναι ΜΜΕ. Η Κομισιόν θα πρέπει να επιδιώξει μια συμφωνία που όλοι θα κερδίσουν εντό τη διαπραγματική εντολή και να σεβαστεί του όρου του Ιουλίου για τη σύναψη τη συμφωνία. Και θα πρέπει να αντιταχθούμε σε οποιασδήποτε προσπάθεια τη Αμερική να συμπεριληφθεί η Γεωργία, όπω είπε ο JFK. Δεν θα πρέπει να διαπραγματεύσουμε το φόβο, ούτε να φοβόμαστε να διαπραγματευτούμε. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε αν έχουμε το πολιτικό κουράγιο, κυρία Ζαντό. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Κόφοντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Το αν θα πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά διαπραγματεύσει είναι νομίζω σαφές για όλους ότι η κυβέρνηση Τραμπ υπονομεύει ε, όλα όσα πιστεύουμε εμείς και οι Αμερικανοί. Και είχα πάει και στις είπαμε μια αντιπροσωπή και υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί μας στο Κογκρέσο που έχουν τελείως διαφορετική άποψη από τον Τραμπ, ο Ρος και την λυπη κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να συζητάμε με ανθρώπους που δεν συμφωνούμε, που υπονομεύουν το κράτος δικαίου στο εμπόριο, που υπονομεύουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Θα πρέπει να το κάνουμε, γιατί η Ευρώπη είναι μια υπερδύναμη εμπορίου. Εμείς έχουμε τον ηγετικό ρόλο. Και βεβαίως ποτέ δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε συμφωνία πριν αρθούν οι μονομερείς δασμοί. Οπότε, εάν αποκατασταθεί βεβαίω ε, κάπου το κρατσουκέο να το δεχτούμε. Αλλά όχι υποπίεση. Κύριε Κόφοντ, μπλε κάρτα τον κύριο Έθριντς Ναι, όχι. Ναι, παρακαλώ. Κύριε ναι. Μπλε κάρτα είχατε ζητήσει. Ευχαριστώ που δεχτήκατε την ερώτηση. Ε, θέλω να μου διευκρινίσετε. Αυτά τα οποία είπατε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερδύναμη, όπως είπατε, δεν θα πρέπει να συνομιλεί με μια κυβέρνηση με την οποία διαφωνεί ε, ακόμα και αν αυτή την χάνει να είναι η πραγματική υπερδύναμη είπα και προτιμάτε να μιλάτε με την αντιπολίτευση αντί με αυτούς που μπορούν να συνάψουν συμφωνία. Εντάξει, καταλαβαίνω τι είναι να έχετε κυβέρνηση που δεν σας αρέσει, το ξέρω, αλλά οπωσδήποτε, εάν μιλάμε για ζητήματα που επηρεάζουν όλες τις χώρες μας, θα πρέπει να συζητάμε το εμπόριο για τις δουλειές και την απασχόληση κτλ. Κύριε Κόφοντ, ε, με παρεξηγήσατε. Μπορούμε να μιλήσουμε με την Αμερικανική κυβέρνηση παρόλες τις διαφορές μας. Γιατί οι ΥΠΑ είναι πολύ ευρύτερες από την τρέχουσα κυβέρνηση. Είναι το Κογκρέσο, όπου πολλοί άνθρωποι διαφωνούν εντόνως με την εμπορική πολιτική του Τραμπ. Και ε, σας είπα ότι είμαστε μια εμπορική υπερδύναμη. Εμείς τηρούμε το κράτος και στο θέμα αυτό. Θέλουμε να ενσωματώσουμε την κλιματική αλλαγή στα ζητήματα εμπορίου και μπορούμε να μιλούμε από θέση ισχύω. Δεν είμαστε αδύναμοι για να μην μιλάμε με ανθρώπου που διαφωνούμε. Σα ευχαριστώ. Ντορνάνο για ένα λεπτό. Euh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ορίστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να ξανανοίξει τι διαπραγματεύσει για να περάσει μια εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ Ωστόσο, οι λαοί απορρίπτουν ε, κάθετα αυτές ε, τις συμφωνίες που τους ε, φτωχαίνουν. Η συμφωνία που προβλέπεται βρίσκεται σε αδιέξοδο από την εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ. Ε, αντί να σημειώσετε αυτή την αποτυχία, οι τεχνοκράτες προσπαθούν να βρουν τεχνάσματα να την αντικαταστήσουν. Σήμερα το βλέπουμε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα το θετικό να παραμένουμε από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πώς να πιστέψουμε ότι η Γεωργία πραγματικά θα αποκλειστεί όταν ο κύριος Γιούνκερ ήδη δέχτηκε και να αυξήσει τις εισαγωγές σόγιας από την Αμερική για να μπορεί να πουλήσει γερμανικά αυτοκίνητα. Θα πρέπει να έχουμε ένα άλλο πιο κοινωνικό, βιώσιμο μοντέλο που να σέβεται τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Κάθε μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει ότι ένα μόνο πρέπει να ε, κάνει, να βγει από αυτήν την κατάσταση για να τα καταφέρει. Αυτοί ήταν οι ομιλητές που μας είχαν δώσει οι ομάδες και περνάμε στη διαδικασία και Έχω μια μεγάλη παράκληση. Δέκα συναδελφοί έχουν ζητήσει τον λόγο. Να σας πω πως για να μιλήσετε όλοι πρέπει να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν και οι δέκα. Κύριος Γιαστρουκεύσκη, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Έχουμε συμφωνία με την Ιαπωνία Προσφάτως συγκρίναμε μια συμφωνία με το Αφγανιστάν. Αλλά τώρα θέλουμε να απορρίψουμε συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Η άκρα αριστερά θεωρεί ότι πρέπει να απορρίψουμε τη διαπραγματευσή. Γιατί, γιατί δεν τους αρέσει ο Τραμπ. Ε, αρέσει στους Αμερικάνους. εσύ θεωρείτε τι, ότι ήταν λάθος οι αμερικανικές εκλογές. Ε, το Brexit ήταν λάθος. Εντάξει, και λάθη αλλά η ΕΠΑ είναι ένας σοβαρός εταίρος ε, και έχουμε δεσμούς ε, αμυντικούς παραδείγματο χάρη πρέπει να είναι λοιπόν στρατηγικός εταίρος και στο εμπόριο και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το εμπόριο με τη ΕΠΑ σας ευχαριστώ κυρία Ροντρίγκες Πινέρο για ένα λεπτό Κυρία Επιτροπέ, υπερασπίζω τι διεθντικέ σχέσει και το διάλογο ως μηχανισμό να επιληθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όμω ειλικρινά δεν πιστεύω ότι τώρα πληρούνται οι προποθέσει να διαπραγματευτούμε εμπορική συμφωνία με τι ΗΠΑ επί του όρου που έθεσε η Κομισιόν. Νομίζω ότι στην πολιτική το πιο σημαντικό είναι η συνοχή μεταξύ λόγων και πράξεων. Και θέλω να απευθυνθώ στου νέου που είναι εδώ, που είναι δεσμευμένοι για την ε, μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και ζητούν δράση από τους πολιτικούς για το μέλλον τους. Και εμείς ε, αν εγκρίνουμε στο Κοινοβούλιο και αν υπήρχε δέσμευση από τα Ευρωπαϊκά Όργανα την κλιματική αλλαγή, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ε, μία εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με αυτούς γιατί δεν θεωρείται ένας εταίρος αξιόπιστος. Μας έχει βάλει κάποιους δεσμούς αδικαιολόγητους και ε, μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί την ασφαλειά τους. Όμως αυτή δεν είναι η όρια για να ξεκινήσουμε ένα διάλογο ε, όπως θα έπρεπε να είναι στο μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμασιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπα, είναι ο μεγαλύτερο παγκόσμιο εταίρος μας. Άρα θα πρέπει να αναμένουμε μακροχρόνιες αμοιβέ ε, δεσμεύσει για να αναπτύξουμε τι εμπορικέ μα σχέσει. Χαίρομαι που βλέπω αυτό το νέο κεφάλαιο να ξεκινάει μετά την κατάρρευση τη TTIP. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην επαναλάβουμε τα παλιά λάθη και αυτή η νέα συμφωνία θα καλύψει όλε τι βιομηχανίε. Δεν πρέπει να είμαστε σκλάβοι ε, στην εναρμόνιση των προτύπων παραγωγής. Θα πρέπει να έχουμε την αμοιβαία αναγνώριση νέων προτύπων, ιδιαίτερα ε, στην επισήμανση των προϊόντων. Πιστεύω ότι οι διαπραγματευτέ μας δεν πρέπει να φέρουν στο τραπέζι οποιασδήποτε ε, προκαταλήψεις για την κυβέρνηση Τραμπ. Αν συνεχίσουμε να στέλνουμε πολιτικά μηνύματα για την ε, διακυβέρνηση του Τραμπ, Αντί να εστιάζουμε την προσοχή μας ε, στην επιχείρηση, θα αποτύχουμε. Το θέμα είναι, θα, θα ξαναδοκιμάσουμε και πότε. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε σοφοί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θέλω να εκφράσω ότι συμφωνώ με αυτές τις διαπραγματικές εντολές για τρεις λόγους. Η οικονομία μας θα αυξηθεί περισσότερο τα επόμενα έτη χάρη ε, από τις εξαγωγές μας στο εξωτερικό. Καταρχήν, ε, το, είναι υποχρεωτικό να προετοιμαστούμε για την κατάσταση για την ευρωπαϊκή οικονομία και προκειμένου μικρέ και μισέ επιχειρήσει να μπορούν να λειτουργήσουν σε κοινή τη χώρα. Δεύτερον, οι συμφωνίε αυτέ είναι η μόνη οδό να υπερασπίσουμε τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μας πρότυπα και να τα διευρύνουμε. Τρίτον, αυτό δεν είναι μεμονωμένη πράξη. Η Ευρώπη έχει απαντήσει στην απειλή του νεοπροστατευτισμού και των εμπορικών πολέμων με την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών όπως αυτή με την Ιαπωνία και αυτές που διαπραγματευόμαστε με ε, άλλους και υποχρεώνει τους λοιπούς να κινηθούν ε, εδώ τα άλογη, τα κενά λόγια και η στετεστερώνη αρέσει στον Τραμπ ε, και κρύβει την, ε, σε αυτά την αποτυχία των συνταγών που υπερασπίζει. Όμως η κυρία Μάλστρομ ε, πέρα από το βιογραφικό της έχει και η ικανότητα να διαπραγματευτεί. Γι' αυτό η πολιτική, η θεαματική που γίνεται θέαμα δεν θα καταφέρει να σας διώξει από το τραπέζι. Και διακόπτε το μικρόφωνο της Κυρία Σκότ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, το να μπούμε σε εμπορικές διαπραγματεύσεις με ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι θα συνεργήσουμε και εμείς στην διάλυση των μέσων του διεθνούς εμπορίου. Θα καταστεί έτσι παροδία το εμπόριο για όλους και θα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο μιας πολιτικής η οποία θα βασίζεται σε κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη με το διακυβερνητικό πάνελ για την κλιματική αλλαγή που λέει ότι έχουμε μόνο 12 χρόνια για το κλίμα, δεν μπορούμε να ανοίξουμε διαπραγματεύσεις με την χώρα η οποία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ε, παραγωγός εκπομπών και αποφεύγει τις κλιματικές δεσμεύσεις. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερους εμπορικούς όρους ένα χρόνο μετά τους τιμωρητικούς δασμούς στην βιομηχανία μας, ενώ την δικιά τους ε, τη χαλιβουργία δεν φροντίζουν να την προσαρμόσουν στη Συμφωνία των Παρισίων. Πρέπει να υπερασπίσουμε την βιομηχανία και τους Ευρωπαίους εργαζόμενους και να πάμε προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Σας ευχαριστώ η κυρία Νταμάτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί δεν θα σας επιτρέψουμε ε, να παρακάμψετε τη δική μας άποψη και των ε, λαών. Πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ που αποτελεί ένα είδος καμουφλαρισμένης συμφωνίας που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των περιβάλλων, επιτρέπει ε, να μπουν από τις Ηνωμένε Πολιτείε προϊόντα γεωργικά και αλίας. Θα ήταν πραγματικά παράλογο και μάλιστα θα ακόμη περισσότερο όλο τον τομέα της ελίας μας και, ε, δεν, και θα ε, έδινε, ε, ούτε θα έδινε ε, χαμηλά συχθείς στους καταναλωτές. Οι εμπορικές συμφωνίες, ναι, πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να υπερασπίσουμε καταρχήν το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και θα πρέπει να δημιουργηθούν αγορές ενδιαφέρουσες και για τους παραγωγούς μας. Όσες φορές και να ρωτήσετε, η δική μας απάντηση θα είναι πάντοτε όχι σε μια νέα TTIP. ένα λεπτό. Η έναξη των διαπραγματεύσεων στοχεύει στο να αποφευχθεί η κλιμάκωση των ε, εντάσεων ανάμεσα σε ΕΕ και τη ΕΠΑ φτάνει οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν, οι δεν θα επιβάλλουν δασμούς στα αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Το 85% της παραγωγής αυτοκινήτων της Πολωνίας ε, ε, αποτέλεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Άρα, είναι προς το συμφέρον μας της Πολωνίας να αποφύγουμε οποιουσδήποτε νέους δασμούς. Επίσης, Έχουμε κλάδους ε, της οικονομίας που είναι εντατική από πλευράς ενέργειας και ε, μιλάμε και για τους κανονισμούς επίσης σε αυτόν τον τομέα, ανάμεσα της ΙΠΑ και την Πολωνία. Η εισαγωγή, για παράδειγμα, υγροποιημένου φυσικού αέριου θα ήταν καλύτερο για μας, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Κύριε Γκραπίνη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σίγουρα έχουμε πολλού λόγου να είμαστε θυμωμένοι με την κυβέρνηση Τραμπ. Εγώ προσωπικά ε, αγωνίστηκα στη TTIP και είχα καταθέσει πολλέ τροπολογίε και κατέπεσε η TTIP. Η σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση όμω με τη ΣΥΠΑ δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε από κοινού τι κερδίσουμε και τι χάνουμε. Εγώ πιστεύω στην Επίτροπο και πιστεύω ότι για μια περιορισμένη εντολή θα πνέξουν οι διαπραγματεύσει. Δεν χάνονται γίνονται παρά οι μάχε που δεν έχουν ξεκινήσει ποτέ, έλεγε ο Άντε, Θα πρέπει να πούμε ότι χρειαζόμαστε την σταξιολόγηση συμμόρφωση, χρειαζόμαστε πρότυπα προϊόντων που είναι αναγνωρισμένα. Χρειάζεται να μην μα επιβάλλουν μονομερού δασμού σε ορισμένα προϊόντα. Και νομίζω ότι εσεί μπορείτε να ε, υλοποιήσετε ε, αυτό το έργο. Ε, να μην έχουμε με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τη ΣΥΠΑ, να μην έχουμε με κανέναν σχέση και με ποιον θα αναπτύξουμε την ενιαία αγορά. Εγώ ελπίζω να περάσουν αυτές οι διαπραγματευτικές εντολές. Ευχαριστώ. Κύριε ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, ονειρεύομαι μια Ευρώπη, Ευρώπη όπου θα έχουμε μια συνοχή της κοινωνικής, αγροτικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Επίτροπε, εξηγήστε μας το συμφέρον της αύξησης των εισαγωγών σόγιας αμερικανικής στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αντί να αυξήσουμε την παραγωγή των ε, φυτικών πρωτεϊνών. Γιατί να ε, θυσιάσουμε την γεωργία μέσα σε όλες αυτές τις ε, συμφωνίες που προτείνεται. Οι μασικές εισαγωγές ε, ε, της σόγιας που είναι εναντίον της Συμφωνίας των Παρισιών. Εσείς ε, που προέρχεστε από μια πολύ όμορφη χώρα θα μπορείτε να βάλετε σε συνοχή αυτή την πολιτική με την αναγκαία μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη που είναι επιτακτική. Ευχαριστώ. Η κυρία για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, έχω την εντύπωση ότι όλα εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν πρόκειται για την απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών. Τα επιχείρηματά σα, ναι, μπορούμε να τα ακούσουμε και ε, να λέμε ότι συνάπτουμε συμφωνίε με φίλες χώρε που συμμερίζονται τι αξίε και του κανόνε μα. Πείτε μου, σε τι ο κύριο Τραμπ και η κυβέρνησή του μοιράζονται τις αξίες μας, τις κλιματικές μας αξίες, ε, αποφάσισε να βγει από τις διαπραγματεύσεις και από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων της COP21 τις αξίες ε, διεθνές εμπόριο. Αποφάσισε ο κ. Τράπ να μην σεβαστεί τους κανόνες του ΠΟΕ. Εσείς που υπερασπίζεται τους κανόνες του ΠΟΕ. Γιατί λοιπόν θέλετε να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ αυτή η ίδια κυβέρνηση δεν σέβεται τους κανόνες που εσείς ζητάτε να σεβαστεί. Σας ρωτώ λοιπόν, ποιο είναι το ένα και μόνο επιχείρημα που έχετε που θα μας επιτρέψει να πείτε, να πούμε ότι είστε σε θέση να αλλάξετε την πολιτική αυτή που δεν σέβεται την Ευρώπη. Ε, αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ σήμερα. Δεν πιστεύω ότι είναι καλό σήμερα να δώσουμε την εντολή που προτείνεται στο Συμβούλιο. Ήταν η τοποθετήση στο πλαίσιο του Τον λόγο τώρα έχει κυρία Επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η συμφωνία που ο κύριο Γιούγκερ σύναψε τον Ιούλιο με τον Πρόεδρο Τραμπ ήταν ε, παρά τις διαφωνίες μας σε κάποιους ε, τομείς να προσπαθήσει να βρούμε τρόπους και χώρους συνεργασίας. Μιλήσαμε για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Υπάρχει επιθυμία από πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε ε, για αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και οι Αμερικανικοί συμφώνησαν να το διευκολύνουν αυτό. Είναι απόφαση κάθε κράτου μέλου και των εταιριών. Δεν είναι η Κομισιόν που αγοράζει το φυσικό αέριο. Η αύξηση ε, τη σόγια και πάλι είναι αποτέλεσμα των αγορών. Η Επιτροπή δεν αγοράζει σόγια και δεν τι αποθηκεύει στον Περλεμόν. Είναι πολιτική τη αγορά, είχε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Συμφωνήσαμε να αποδεχτούμε το σχέδιο αηφορία τη Αμερική ε, με πλήρη συμμόρφωση προ την οδηγία. Συμφωνήσαμε ότι θα συνεργαστούμε για να μεταρρυθμίσουμε ε, την ε, ΠΟΕΜ. Υπήρχε διαφωνίε, αλλά έχουμε μία διαδικασία όπου συνεργαζόμαστε με του Αμερικανού και του Ιάπωνε για να καταγράψουμε νέου κανόνε στον ΠΟΕ για να αντισταθμίσουμε ανταγωνισμό από την Κίνα. Επίση, κανονιστική ε, διαδικασία στον τομέα των τροφίμων με πλήρη σεβασμό προς τα προστατευτικά συστήματά μας. Και επίσης συμφωνήσαμε ότι θα επιστήσουμε διαπραγματεύσεις σε δύο περιορισμένες συμφωνίες ε, τη συμμόρφωση της αξιοπιστίας, αξιολόγηση της και δεύτερον ε, στα ε, στους δασμούς για τα βιομηχανικά αγαθά. Και εδώ ζητάμε την άποψή σας εδώ. Ε, στην εντολή υπάρχουν σαφείς όροι. Δεν μπορούμε να συνάψουμε οτιδήποτε εάν οι δασμοί ε, του χάλιβα και του αλουμίνιου δεν αρθούν. Δεν θα υπάρχουν επιπροσθετοί δασμοί στο κεφαλαίο 232, στα αυτοκίνητα επίσης. Στη σειρά αυτών των διαπραγματεύσεων θα κάνουμε μια εξωτερική μελέτη ε, αντικτύπου των επιπτώσεων της ειφορίας και έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Είναι ξεκάθαρο αυτή την εντολή και ε, με το να την αποδεχτείτε θα πείτε ότι δεν περιλαμβάνεται η γεωργία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι μια περιορισμένη συμφωνία. Ε, συμπτάμε για τα ε, βιομηχανικά αγαθά ε, συμπεριλαμβανομένη τη αλίας και των αυτοκινήτων. Και τα ποσά δεν είναι αμεληταία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεν είναι μια πλήρη συμφωνία ελευθερών συνάλλαγων. Δεν αφαιρείται η TTIP. Η TTIP είναι στο ψυκτικό θάλαμο. Δεν κατέστη δυνατό να την ακολουθήσουμε υπό ε, ε κυβέρνηση Ομπάμα και δεν προβλέπεται ούτε και τώρα. Και φυσικά το έχετε αναφέρει κι εσείς, ε, διότι οι ΗΠΑ έχουν αποσυρθεί από την Συμφωνία των Παρισίων. Υπάρχουν, όπως είπα, αρκετές διαφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά η είπα ο λαός, οι εκλεγμένες συνελεύσει στο έθνος είναι φίλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε κάθε συμφέρον να προσπαθούμε να βρούμε το μη συνεργασίας, το μη συνομιλίας και διαλόγου μαζί τους. Και αυτή είναι η βούληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ομόφωνα επίσης. Και γι' αυτό ζητάμε να συμφωνήσετε για αυτή τις δύο διαφορετικές εντολές ε, και ελπίζω ότι θα υπερψηφίσετε επίσης αύριο αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπή, κύριε Βέσοβιτς, να σας πω ότι δεν μπόρεσα να σας δώσω τον λόγο γιατί είχατε πάρει ε, μπλε κάρτα. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να σας δώσω δύο φορές τον λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση έχουν υποβληθεί μια σειρά ε, ψηφισμάτων ε, της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση. Η ψηφοφορία είναι αύριο. Επόμενο θέμα. Έχουμε την κοινή συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την Οικονομική Πολιτική και τον συντονισμό της. Έκθεση Φαντεν Κέντελάρε. Με συγχωρείτε αν δεν πρόφερα σωστά το όνομά σας. Ετήσια έκθεση 2019 και έκθεση Χάρκιν, επίσης Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό της Οικονομικής Πολιτικής, Απασχόληση και Κοινωνικές Πτυχές στην ετήσια έκθεση ανάπτυξης 2019. Πρώτα απ' όλα, τον λόγο έχει ο κύριος Φαντεκέντελάρη. για τέσσερα λεπτά. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, αγαπητοί Επίτροποι, συνάδελφοι. Οι συζητήσει για το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι πολύ πολιτικά φορτισμένες και όσο πλησιάζουν εκλογές ε, η κατάσταση αυτή θα επιδεινώνεται τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε είναι ακριβώς αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν πολιτικά. Ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας μας δηλαδή, ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις, ποιες προτεραιότητες έχουμε και κυρίως πώς θα φροντίσουμε να μεταδώσουμε το κράτος δικαίου που έχουμε στα παιδιά μας και το κράτος πρόνοιας. Άλλοι ζητάνε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, άλλοι ζητάνε περισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία και άλλοι πάλι ζητάνε να στηρίξουμε πράσινα έργα. Ως χριστιανοδημοκράτης ε, θεωρώ ότι η καλύτερη πορεία είναι ο συνδυασμός όλων αυτών. Με μισές αλήθειες και εύκολες λύσεις δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει λοιπόν για αυτούς και για τα παιδιά μας να τους πούμε ολόκληρη την αλήθεια. Συμπτωματικά είναι εδώ πέρα ο γιος μου, ε, δύο ετών, σήμερα και αύριο, και γι' αυτόν βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Θέλω στο μέλλον ε, το κράτος πρόνοιας ε, το οποίο φροντίζει αυτόν ε, και τους συγγενείς του όσο και αν δύσκολο φαίνεται να μπορεί να τον φροντίζει αν αρρωστήσει και βεβαίως όταν θα έχει δουλέψει σε όλο και τη ζωή να του δώσει και μια σύνταξη. Αυτό το μέλλον η κληρονομία 10 ετιών ε, είναι αυτό το οποίο είναι το διακύβημα. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, η γύρανση είναι μια πολύ σημαντική δημογραφική εξέλιξη του 21ου αιώνα. Από μόνη της είναι μια τεράστια εξέλιξη, αλλά βεβαίως σημαίνει και δύο μεγάλες προκλήσεις. Πρώτον, το κόστος των συντάξεων της υγείας και της φροντίδας των ηλικιωμένων, τα οποία θα αυξηθούν τις επόμενες δεκαετίες και θα πιέσουν τα δημόσια οικονομικά. Και δεύτερον, γύρανση σημαίνει ότι θα έχουμε αναλογικά, αναλογικά με λιγότερους εργαζόμενους οι οποίοι θα πρέπει να υπομιστούν αυτό το κόστος και πάλι λοιπόν πίεση στα δημόσια οικονομικά. Πρέπει λοιπόν να παρέμβουμε σε τρία μέτωπα. Πρέπει και να επενδύσουμε και να υπάρξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να έχουμε τακτοποιημένους προπολογισμού. Πρώτον, λοιπόν, υγιή δημόσια οικονομικά. Πρέπει να έχουμε αποθέματα τα οποία θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το κόστος της γύρανσης. Περισσότεροι ηλικιωμένοι σημαίνει περισσότεροι συνταξιούχοι, περισσότερο κόστος για την υγεία. Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε. Αλλιώς θα πασάρουμε το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Δεύτερον, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος αυτό και έτσι να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν εύκολα δουλειά και οι εργοδότες βεβαίως να μπορούν να προσλαμβάνουν και να απολύουν ευκολότερα. Οι γονείς μου ήταν μια γενιά η οποία δούλεψε σε ολόκληρη τη ζωή της ε, σε μια επιχείρηση. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα κάνει πιο εύκολη αυτή την μετάβαση. Να έχουμε δηλαδή τους εργαζόμενους οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να είναι ευέλικτοι, να έχουν διαβίου κατάρτιση. Και τέλος, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά την γύρανση, πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον. Όχι μόνο σε ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως είπα, αλλά και στην μελλοντική παραγωγικότητα για να διασφαλίσουμε την οικονομική μας ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση και στις υποδομές. Λογικές επενδύσεις σήμερα σημαίνουν αποδόσεις αύριο. Αυτό πρέπει να κάνουμε με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, μια, ένας μπούσουλας κοινωνικο-οικονομικός, ο οποίος θα μας καθοδηγήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. ευχαριστώ. κυρία Χάρκιν για τέσσερα λεπτά Να ευχαριστήσω καταρχήν τους και συζητητές για την καλή συνεργασία που πιστεύω ότι οδήγησε σε μια ισορροπημένη έκθεση. Υπάρχουν κάποιε τροπολογίε που έχουν υποβληθεί και νομίζω ότι με την εξαίρεση μία μπορώ να τι υποστηρίξω όλε. Δεν αλλάζουν σημαντικά το περιεχόμενο ή το ύφο τη έκθεση, αλλά βελτιώνουν το κείμενο. Καταρχήν, να πω Πόσο σημαντικό είναι για την Επιτροπή Επασχόληση να έχει τη δική τη ξεχωριστή έκθεση για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη, γιατί έχουμε διαφορετική προοπτική από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Είναι συμπληρωματικέ, αλλά έχουν διαφορετική έμφαση. Και αυτή η έκθεση και οι προηγούμενε δύο εκθέσει τη Επιτροπή επασχόληση πιστεύω ότι συνεισφέρουν ε, στην επαναξισορρόπηση τη σημασία